και όλα. Και πολλοί συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους αυτό ακριβώς διεκδικούν ενίσχυση και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Ό,τι αφορά τις α, τροπολογίες, έχουν υποβληθεί τροπολογίες από τις κυρίες Μακοβέη Λάτφορτ και τον κύριο Κυρκόπ. Τροπολογίες που προσθέτουν δύο νέα κριτήρια για την αξιολόγηση. Την ανεξαρτησία και την ταχύτητα των δικαστικών οργάνων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα να πω για να διασκεδάσω τις αμφιβολίες σας ότι συμμερίζομαι και εγώ αυτές τις ανησυχίες και το θέμα είναι αν μπορούμε να εισαγάγουμε νέα κριτήρια με την πρωτοβουλία αυτή στο μηχανισμό αξιολόγησης Σέγγεν. Γιατί η νομική γνωμοδότηση που ζήτησα μου λέει ότι δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βρούμε άλλη ευκαιρία για να προσθέσουμε νέα κριτήρια στα ήδη υπάρχοντα του Σέγγεν. Σε τελική ανάλυση θα μπορούσαμε με τέτοιου είδους ανησυχίες να τις ε, συμπεριλάβουμε μόνο στο μέτρο που έχουν συνέπειες συγκεκριμένε στα κριτήρια, στα υπάρχοντα κριτήρια Σέγγεν. Αλλά για την πρόταση ενός μηχανισμού, στην πρόταση ενός μηχανισμού αξιολόγησης δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το κεκτημένο Σέγγεν. Γι' αυτό και θα προτείνω μια συμβαστική λύση που θα ε, ασθενίζεται τις και θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των ε, Κίρκοπ, Μακοβέη και Λάτφορτ, αλλά θα πληρεί και τις νομικές προϋποθέσεις και τους νομικούς περιορισμούς που μας δεσμεύουν. Και στη, στο μέλλον, όταν εξετάσουμε πρόταση αναθεώρησης του κεκτημένου Σέγγεν, εκεί είμαι πρόθυμος να συνυπογράψω και με αυτούς τους συναδέλφους και με άλλους πρόταση για την διεύρυνση των κριτηρίων που προβλέπονται στο κεκτημένο Σέγγεν. Σε ό,τι φορά τις τροπολογίες κυρίας Μακοβέη για το ρόλο της Europol, θα ήθελα να πω ότι έχω την αίσθηση ότι ιδιαίτερα για θέματα ανάλυσης κινδύνου μπορεί να γίνει δεκτή η πρότασή της. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τροποποιηθεί η διατύπωση αυτή. Προκειμένου να ανταποκρίνεται στα υπάρχοντα κριτήρια του Σέγγεν, δηλαδή καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, λαθρεμπορίου όπλων και δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα μέσω της κυρίας Βέμπερ να διαμηνήσω στην κυρία Λάτφορτ ότι σε μια δική μου τροπολογία ήδη είχα καλύψει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας προκειμένου να, να λάβω υπόψη την μερική του συμμετοχή στο Σέγγεν. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την κυρία Λάτφορτ. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις τροπολογίες των Μαρινέσκου, Εντσίου, Νέλτσεβα, Παπα-Νικολάου και Κιγκαγκόντς. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες της ΓΚΟΕ, θα συνεννοηθώ με τους συντάκτες τροπολογιών για να καταλάβω ποιο είναι ο στόχο τους, για να δω πόσους μπορώ να δεχτώ. Και αντίστοιχη επιφύλαξη έχω και μία τροπολογία του κυρίου Λαμπρινίδη. Θα ήθελα μέσω ημών, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσω από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Λόπες Ακυλάρ, να υποβάλλει προς την νομική υπηρεσία μία ερώτηση ως προς τη θέση της νομικής υπηρεσίας για τη νομική βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαμάχη μεταξύ δύο νομικών υπηρεσιών. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υποστηρίζει ε, την ε, υπάρχουσα νομική βάση ως σωστή συμφωνώ, αλλά έχουμε και μια πρωτοβουλία πολλών χωρών μελών που φαίνεται ότι στηρίζονται σε μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και που τάσσονται υπέρ μιας διαφορετικής νομικής βάσης. Έχουμε μια πραγματική διαμάχη μεταξύ των νομικών υπηρεσιών για τη νομική βάση. Είναι χρήσιμο αυτή την άποψη να ζητήσουμε τη γνωμοδότηση και της δικής μας νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αποφανθεί και αυτή η νομική υπηρεσία για το ποια νομική βάση κρίνει δόκιμη. Τη βάση που προτείνει η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη νομική βάση που προτείνει η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Καρλός. Βλέπω ότι ανακύπτουν όλο και νέα ζητήματα που χρήζουν διευκρίνησης και είναι νομικής υφής. Τώρα θα το λόγο στην κυρία Χουσάρ, την εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. bizottságot a tanácsban zajló tárgyalások állása. Fejfele? Ne. Nagy jelentőségű. Sorry, Mrs. President, I have no translation in Portuguese. Ο εισηγητής Κουέλου αναφέρει ότι δεν έχει διερμηνία προς τα πορτογαλικά. From Okay. I, It, it's soft. Thank you so much. Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω εξ ονόματος του Συμβουλίου για την κατάσταση πραγμάτων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτή η αξιολόγηση του κεκτημένου του Σέγγεν έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτού του καθεστώτος. Η Ουγγρική Προεδρία κατέστησε αυτό το θέμα μία από τις προτεραιότητες της. Είπαμε με τον κύριο Κουέλιο ότι χρειάζονται περισσότερες ε, κυρώσεις και σοβαρότερες κυρώσεις για αυτούς που δεν ε, ε, εφαρμόζουν το κεκτημένο του Σέγγεν. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν ε, ενισχυμένο ρόλο και θέλουμε την καλύτερη εφαρμογή του όλου καθεστώτος έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις. Χρειάζεται καλύτερη κατανομή εργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να αναφέρω στους βουλευτές ότι η επιλογή της νομικής βάσης θα έχει επιπτώσει στην διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, αλλά το Συμβούλιο θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία ανεξάρτητα από τη νομική βάση που θα επικρατήσει. Στα πλαίσια του Συμβουλίου, η πλειοψηφία των κρατών μελών θεωρεί, όπως αναφέρει η νομική υπηρεσία, ε, θεωρεί ότι η αξιολόγηση του κεκτημένου του Σέγγεν δεν απορρέει από τη νομική βάση όπως όριζε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ε, Ουγγρική Προεδρία δέχτηκε αυτή τη γνωμοδότηση της νομικής ε, υπηρεσίας. Η Προεδρία δεν κρίνει σκόπιμο να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτή την πρόταση, διότι η τελική έκβαση εξαρτάται εμπολής από την πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο ως προς το μέλλον του καθεστώτος του Σέγγεν. Οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά από την λήξη της πολιτικής συζήτησης είναι γεγονός ότι το σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να ενισχυθεί και τα βήματα, τα μελλοντικά μας βήματα θα εξαρτηθούν από τις στρατηγικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μόνικα Μασάμπα. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πολλές είναι ενδιαφέρουσες ιδέες στις τροπολογίες που κατατέθηκαν και θα ήθελα να απαντήσω έτσι με γενικό τρόπο στις διάφορες κατηγορίες τροπολογιών. Βεβαίως η τεχνική προσαρμογή είναι θέμα της επιτροπολογίας και βεβαίως προφανές. Ε, αλλά Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες για να λειτουργούν καλύτερα οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, να συμμετέχουν ενδεχομένω περισσότερο και τα κράτη-μέλη. Εντάξει, προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων, ανέφερε την Ευρωπόλη ο εισηγητής. Βεβαίως υπάρχει χώρος να συμμετέχει και η Ευρωπόλ και αυτό αντανακλάται στην πρόταση, αλλά θα πρέπει πάντα να κοιτάμε την εντολή και το κεκτημένο που θα πρέπει να αξιολογείται γιατί βεβαίως υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, αλλά έχουν ο καθένα την εντολή του στην Ένωση και αυτό θα πρέπει πάντα να το προσέχουμε. Να δούμε ε, σε ποιο σημείο και μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξη των διαφόρων οργανισμών. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που ζητούν να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδατε ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δείχνει κάθε ειλικρίνεια και διαφάνεια και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Ωστόσο κάποιες τροπολογίες νομίζω είναι υπερβολικές για την καθημερινή δουλειά της αξιολόγησης του Σέγγεν. Δεν είμαι βέβαιη αν θα θέλατε όλοι να λαμβάνετε τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ή στα προγράμματα δράσης, πώς ε, εφαρμόζονται γιατί εσείς έχετε άλλη δουλειά ως θεσμικό όργανο. Δεν μπορεί να είστε τόσο πολύ στην καθημερινότητα ε, της αξιολόγησης του κεκτημένου Σέγγιν. Βεβαίως παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα που ε, εξαρτώνται από την πολιτική καθοδήγηση που θα πρέπει να λάβουμε. Το ένα είναι η εισαγωγή κυρώσεων και θα ήθελα να αναφέρω ε, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 4 Μαΐου, εάν και κατά πόσο σε έκτακτες περιστάσεις μπορούν να επανέλθουν οι έλεγχοι στα σύνορα. Αυτό είναι θέμα που θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δούμε πώς θα μας καθοδηγήσει. Για ε, το πρώτο και το δεύτερο τμήμα της εντολής, ο κύριος Κοέγιο ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε διπλά ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται και ο κανονισμός για το πρώτο τμήμα της ε, εντολής πριν την άρση των ελέγχων στα σύνορα, αλλά αυτό το θα το δούμε στο τέλος ε, της ε, προσχώρησης στο Σέγγεν των μελλοντικών διευρύσεων. Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, συμφωνώ με τον κύριο Κοέλιο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να δούμε Ποια είναι η βάση του κεκτημένου που αξιολογείται και ελέγχεται. Είναι το Σέγγεν και το κεκτημένο του Σέγγεν. Αν είναι εντάξει μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω, αλλά πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι η συγκριτική αξιολόγηση, τα ορόσημα που έχουμε και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσει και για το πεδίο εφαρμογή. Και ένα τελευταίο, χωρί να είναι λιγότερο σημαντικό, η επέκταση προ ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλανδία. Έχω εξηγήσει σε προηγούμενε συνεδριάσει ότι η, ο, όχι ακριβώς αποκλεισμό, η εξαίρεση για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία είναι θέμα νομικής βάσης. Καταλαβαίνω όμως και τα σχόλια που γίνονται ότι δεν είναι δυνατόν να αποφεύγουν, να γλιτώνουν εντό εισαγωγικών την ε, αξιολόγηση του Ηνωμένου Βασίλειου και Ιρλανδία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Έντσου, Τζανόκα, Βέμπερ, Ναντέλτσεβα, Μακοβέη. Uh, uh, Μάλιστα. Ο κύριος Έντσου. Καταρχήν, για άλλη μια φορά, θα ήθελα να τονίσω τον επαγγελματισμό του κυρίου Κοέλιος προς την ε, προετοιμασία αυτής της έκθεσης και την ανάλυση των ανακοινώσεων της Κομισιόν. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των τροπολογιών συνεισφέρουν θετικά για την βελτίωση του μηχανισμού αξιολόγησης του κεκτημένου του Σέγγεν. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διαφάνεια καταρχήν, λαμβάνοντας υπόψη την, ε, ε, τα αρνητικά προηγούμενα. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε την ε, αξιολόγηση όλες τις φάσεις της. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα και νομίζω ότι οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν αποτελούν μία πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω και το Συμβούλιο να συμφωνήσει με την αρχή ε, ε, διαφάνειας, όπως ορίζει το Κοινοβούλιο. Σε σχέση με τις επισκέψεις των ευρωπαϊκών οργανισμών, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επισκέψεις αυτών των οργανισμών, όπως της Frontex, της Europol, του Ευρωπαίου Επόπτη και ούτω καθεξής επιτόπου. Ε, όπως ε, γνωρίζουμε, μετά από επισκέψεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ευρωβουλευτές σε αυτές τις επισκέψεις ως προς τις αναλύσεις ε, κινδύνων οι τροπολογίες ως προς αυτό το θέμα αφορούν την ενιαία ανάλυση κινδύνου την οποία αναλαμβάνει η Frontex καθώς και οι συστάσεις από άλλους οργανισμούς, δηλαδή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, Frontex και ούτω καθεξής ως πως διαφοροποιημένους, ε, διαφοροποιημένες αναλύσεις κινδύνου από άλλους οργανισμούς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγχυση. Θα ήθελα να θέσω και ένα ζήτημα σε σχέση με τα επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης ε, που τίθενται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ κρατών μελών αυτό αποτελεί απαράβατο όρο για την αξιολόγηση του κεκτημένου. Μπορεί να επέλθει σύγχυση λοιπόν όταν μιλάμε για συνοδευτικά μέτρα επιπροσθέτως των κριτηρίων αξιολόγησης, διότι υπάρχουν ειδικά μέτρα, ειδικέ προδιαγραφές αξιολόγησης ως προς τη διαφθορά και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό θα πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά. Μπορούμε να εισαγάγουμε και επιπρόσθετα κριτήρια, αλλά νομίζω ότι όπως προτείνεται τώρα ε, δεν είναι ικανοποιητικά τα επιπρόσθετα κριτήρια. Θα πρέπει να ε, οριστούν επαρκώς έτσι ώστε οι αξιολογήσεις να είναι σαφείς, διαφανείς και αντικειμενικές. Υπάρχει και μία τροπολογία που συζητήθηκε που αναφέρεται στην περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που δημιουργεί διπλά μέτρα και σταθμά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό και να μην γίνεται αυτή η ειδική αναφορά. Σε σχέση με το μηχανισμό κυρώσεων, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι προτεραιότητες αφορούν τα μέτρα αρρωγής προς ε, το κράτος μέλος που αντιμετωπίζει προβλήματα. Και εάν εμένουν οι δυσχέρειες θα πρέπει να εισαγάγουμε ένα προοδευτικό σύστημα κυρώσεων μέχρι ότου κλείσουμε προσωρινά τα εσωτερικά σύνορα. Αυτό θα πρέπει να γίνει υπό αυστηρές ε, συνθήκες ελέγχου, όπως λέει και ο Κάρλος. Θα πρέπει να ορίσουμε τον χρόνο εφαρμογής των κυρώσεων και εάν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σαφείς. Δεν μπορούμε να ορίσουμε εξαιρέσεις στον κανονισμό ως προς την εφαρμογή του κεκτημένου, διαφορετικά δεν θα επρόκειτο παρά για ένα αρνητικό σύστημα αξιολόγησης, ενώ αυτό μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε το κεκτημένο. Ευχαριστούμε κύριε Έντσου. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο, όχι μόνο για την υποστήριξή του, αλλά για τη θέση του στο Συμβούλιο, γιατί υποστήριξε πολύ καλά την ανάγκη και την απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Εγώ είμαι υπέρ δύο θέσεων του εισηγητού που είναι ε, μείζονος σημασίας και για μας. Θεωρώ ότι η ίδια διαδικασία αξιολόγηση θα πρέπει να ισχύει και για τα κράτη-μέλη του Σέγγεν και για τις υποψήφιες χώρες Σέγγεν. Και συμφωνώ με την πρόταση για τα δεδομένα, για τους διατάξεις και κανόνες προστασίας δεδομένων. Έχουμε και τροπολογία σχετικά. Σε ό,τι αφορά άλλες τροπολογίες θα μπορούσαμε να δεχτούμε πολλές από αυτές, αλλά χρειαζόμαστε προηγουμένως ορισμένες διευκρινήσεις. Για παράδειγμα, ποιος θα πρέπει να συμμετέχει στις ευνίδιες επιτόπιες επισκέψεις. Θα συμμετέχουν στις ομάδες αυτές μόνο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και εμπειρογνώμονες που θα διορίζονται από τα κράτη-μέλη. Φυσικά υπάρχει ανάγκη ανάμειξη και των κρατών μελών, γιατί ο χώρο έγκυση στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πώς όμως θα εξασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, το απόρριτο αυτών των επισκέψεων, ώστε όντω να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που δεν σχετίζονται άμεσα με το κεκτημένο Σέγγεν. Δικαστικέ μεταρρυθμίσει, οργανωμένο έγκλημα, πάταξη διαφθορά. αυτά τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση. Και έχουμε και το θέμα της συνεχούς αξιολόγησης. Μετά την εμπειρία που είχαμε με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία γνωρίζουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα κριτήρια και μάλιστα δεν υπάρχει και σχετική νομική βάση. Βέβαια είναι εύλογε ορισμένες ανησυχίες των χωρών μελών για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση, αλλά πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε σαφείς και προβλέψιμους μηχανισμούς για την δυνατότητα καταμέτρηση οποιοδήποτε νέου κριτηρίου που θα προσθεθεί στον μηχανισμό αξιολόγησης η επανεισαγωγή μεθοριακών ελέγχων θα θεωρηθεί ω κύρωση για τη μη εφαρμογή του κεκτημένου σε ή παραβίαση οποιοδήποτε νέων κριτηρίων. Και εδώ χρειαζόμαστε ένα διαφανές και προβλέψιμο σύστημα. Και τι προβλήματα θα προκύψουν από μια τέτοια επανεισαγωγή. Και για πόσο καιρό θα επανεισαγάγουμε τέτοιους μεθοριακούς ελέγχους, με ποια διαδικασία θα τους επανεισαγάγουμε και πώς θα τις καταργούμε τέτοιους ελέγχους ε, μετά την επανεισαγωγή τους, με ποια διαδικασία. Τέλος, δεν πρόκειται για ερώτηση αλλά για παρατήρηση, για δήλωση. Οι πράσινοι πιστεύουμε ότι μόνο πραγματικές απειλές θα μπορούσαν να είναι λόγος για την επανεισαγωγή τέτοιων ελέγχων στα σύνορα. Και μάλιστα πρέπει να είναι ίστατο μέτρο και να είναι άμεσε αυτέ οι απειλέ και όχι απλώ υποθετικές. Πιστεύουμε ότι πολλοί μετανάστες ή σε άσυλο δεν συνιστούν από μόνο τους απειλή και δεν θα πρέπει να γνωρείτε το κεκτημένο από τους ε, φύλακε των σύνορων. Ελπίζω ότι και στο εγγύς θα καταφέρει ο εισηγητής μας να συντάξει κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που θα λαμβάνουν υπόψη τις επιφυλάξεις μας και θα προβαίνει στις απαραίτητες διευκρινήσεις. Και προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία μαζί του, προκειμένου να έχετε πραγματικά ισχυρή εντολή για τις επόμενες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πέμπερ. ευχαριστώ πρόεδρε. Η όδηση συγγήτριά μας, η Σάρα της δυστυχώ χρειάστηκε να φύγει. Επιστέψει στο Λονδίνο. Είχε άλλη ενήλμένη υποχρέωση. Και θα πω εγώ δύο λόγια εξ της, αλλά και εξ μου. Ε, τώρα βρισκόμαστε σε μια στιγμή που θα τη χαρακτήριζα άκρος ενδιαφέρουσα. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που λέει «Ήθε να ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς». Καμιά φορά είναι πολύ ενδιαφέροντες οι καιροί και για το Σέγγεν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και χαίρομαι που η εισηγητής για αυτά τα θέματα είναι ο κύριος Κάρλος Κοέλιο, γιατί τον εμπιστεύομαι και τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, διαπραγματεύεται. on the, right. Και είμαστε ε, πραγματικά στο σωστό δρόμο. Και έχουμε βρεθεί λοιπόν σε μια χρονική στιγμή όπου τι θέλουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε, να διαφυλάξουμε το Σέγγεν, που είναι τόσο σπουδαίο και εκτιμένο αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών, και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα πρέπει να, επιπλέξουμε, να περιπλέξουμε το Σέγγεν με διάφορα πράγματα που ουσιαστικά θα αποδυναμώσουν, πώς να το πω, θα διαλύσουν ε, την πραγματική δύναμη που έχει αποκτήσει το Σέγγεν. Με αυτό το μηχανισμό αξιολόγησης αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς να προχωρήσουμε με αυτό το δρόμο, να διαφυλάξουμε, να σώσουμε αυτό που έχει επιτευχθεί ήδη στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε να πάμε σε άλλους μηχανισμούς. Ελπίζω ειλικρινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μας φέρει τίποτα επιπλέον. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο εργαζόμαστε σε αυτό το μηχανισμό αξιολόγησης, τον επεξεργαζόμαστε και για τα σύνορα για το Σέγγεν, αυτά αρκούν και καλό είναι να καλύπτουμε ό,τι πρέπει να καλύπτεται σχετικά και τίποτα παραπάνω. Έρχομαι τώρα στις τροπολογίες. Μου κατέθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Προσωπικά, προσωπικά τώρα αυτά δεν τα λέει η Σάρα Λάτφορτ, τα λέω εγώ, γιατί είναι η τροπολογία δικιά της. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις συμβαστικές τροπολογίες μπορεί να αλλάξουμε λίγο το γράμμα, διατηρώντας όμως το πνεύμα της τροπολογίας της. Για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και μηχανισμούς δικαστικής επαλήθευσης, χωρίς αναφορά σε ιδιαίτερες χώρες, δεν είναι σημασία αυτή. δεν έχει σημασία, ούτε είναι και πολύ δίκαιο να κατονομάζουμε χώρες. Διατηρούμε την ουσία αυτού που θέλουμε να πούμε χωρίς να αναφερόμαστε ρητά σε κάποια απόφαση. Από την άλλη, σχετικά με το πώς θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση, ορισμένες τροπολογίες φιλοδοξούν να εντάξουν και άλλα θεσμικά όργανα, άλλου θεσμού αυτό και οργανισμούς, την Ευρωπόλ για παράδειγμα. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί κατά την άποψή μας το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι μπορεί να καλεί την Frontex, την Europol, την Eurojust και όποιον άλλο θεωρεί σκόπιμο ε, να ορίσουν ένα εκπρόσωπο που θα συμμετέχει ως παρατηρητής στην επίσκεψη ε, και θα καλύπτει θέματα των αρμοδιοτήτων φτάνει μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται επιπλέον ε, μηχανισμός γιατί θα αυξηθεί τρομακτικά η ε, γραφειοκρατία του μηχανισμού αξιολόγηση. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι ε, απλός όσο και αποτελεσματικός και να αποδείξουμε ότι κάνουμε τη δουλειά μας ακριβώς για να βεβαιωθούμε ότι η Συμφωνία Σέγγεν παραμένει ισχυρή, είναι ακόμα πιο αποτελεσματική από ό,τι μέχρι σήμερα. Κάτω τα λοιπά, τα πούμε με τον εισηγητή, θα τα διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρενάτα. Βλέπεις Κάρλος, όλοι συμφωνούμε με τη Ρενάτα ότι έχεις κάνει καταπληκτική δουλειά για το Σέγγεν. Η κυρία Ναντέλτσεβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κοέλιο για την έκθεσή του. Είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη. Συμφωνούμε όλοι ότι ε, το κεκτημένο του Σέγγεν και οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα είναι πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρο. Γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε ε, μία από τις πολύ ε, σπουδαίες ε, ελευθερίες και επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν θα πρέπει να χωρίσουμε, θα πρέπει να διαφυλάξουμε ακριβώς την ελεύθερη κυκλοφορία, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Γι' αυτό ζητώ ενισχυμένο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα είναι ο θεματοφύλακας για περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Κάποια κράτη-μέλη μπορεί να δυσκολεύονται να εφαρμόσουν ε, το κεκτημένο του Σέγγεν και είναι πάρα πολύ καλό να τους χορηγείτε βοήθεια για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτό το χώρο του Σέγγεν για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία ε, σημαντικά θέματα και χαίρομαι που τα αναφέρει η έκθεση του κυρίου Κοέλιο. Θέλω να αφαιρθώ συγκεκριμένα στις επισκέψεις και στις επαληθεύσεις πριν, κατά και μετά. Κάθε κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες προδιαγραφές. Έτσι. Και θα πρέπει κάθε κράτος να κρίνεται με τον ίδιο τρόπο. Οι επιτόπου έλεγχοι και επαληθεύσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο ε, αντικειμενικό, αμερόληπτο και να ισχύουν τα ίδια για όλους. Και όχι να βασιζόμαστε σε εικασίες και υποθετικά σενάρια, αλλά σε πραγματικά περιστατικά. Έτσι θα αυξηθεί άλλωστε και η αξιοπιστία του μηχανισμού του Σέγγεν. Κατά τη διάρκεια των επαληθεύσεων, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών, αλλά με πάρα πολύ ε, καλά ορισμένο ρόλο θεσμικό. Ε, Frontex, Europol, Eurojust, δεν ξέρω ποιος θα είναι αρμόδιος και θα έχει οριστεί ε, ως μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων, αλλά με σαφή εντολή για να αποφεύγονται επικαλύψεις αφενός και αφετέρου επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για ορισμένα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καταθέσουν προγράμματα, συντονισμένα όμως, μετά τους ελέγχους. Και εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να αφορούν ε, περισσότερα από ένα κράτος μέλος που έχουν κοινά σύνορα. Λογικό είναι αυτό. Αλλά και πάλι να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία για να μπορούν ταυτόχρονα να δρουν οι χώρες και να είναι πιο αποτελεσματικές. Και τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές ερωτήσεις για την παράγραφο, συγγνώμη, την τροπολογία 87 του εισηγητή για τις κυρώσεις και τη δυνατότητα επανεισαγωγής ελέγχων ε, στα εσωτερικά σύνορα. Τι σημαίνει αυτό παρακαλώ. Ε, και μιλάει για έλεγχους ε, μερικούς ή πλήρης. Πώς γίνεται ο εν μέρη έλεγχος και ποιες είναι οι έκτακτες περιστάσεις. Και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι το εξάμεινο ε, είναι αρκετή χρονική περίοδος και δεν θα ε, παραταθεί. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ ο Κάρλος για την έκθεση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ως συνοδευτικά μέτρα για την αξιολόγηση του μηχανισμού για το κεκτημένο Σέγγεν. Γνωρίζουμε ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σέγγεν. Δεύτερον, χρειάζεται εμπιστοσύνη και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Θα έχω εμπιστοσύνη σε έναν ανώτερο αξιωματούχο μιας άλλης χώρας αν έχω την πεποίθηση ότι δεν είναι διαφθαρμένος. και αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο ορισμένα. Εάν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία βλέπουμε ότι η διαφθορά υπάρχει ε, ίσως σε περισσότερα κράτη από δύο ή τρία. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αυτά. Πιστεύω, έχω την πεποίθηση ότι αυτή είναι η θέση όχι μόνο των Ρουμάνων πολιτών, και το λέω επειδή προέρχομαι από τη Ρουμανία, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς και την αμοιβαία εμπιστοσύνη στο χώρο Σέγγιν. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επίτροπη έλαβε μία απόφαση και πρέπει σε μία ανακοίνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για πρώτη φορά ορίζει μία πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι αυτό το θέμα είναι πρόβλημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αν δείτε την ανακοίνωση καταπολέμησης της διαφθοράς, βλέπετε το κόστος ε, το ετήσιο κόστος φτάνει σε 120 δις ευρώ ετησίως. Και επίσης οι πολίτες, 4 στους πέντε πολίτες θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί μίζον πρόβλημα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 83 της συνθήκης που θεωρεί ότι πρόκειται ότι η διαφθορά είναι ε, ένα σοβαρό αδίκημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτακτικά. Στην τροπολογία 1, ως προς την αιτιολογική σκέψη 1, μιλάμε για αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία είναι ε, αναπόσπαστο στοιχείο για την ε, συνεργασία. Μιλάμε για ε, μέτρα που αφορούν τις, ε, τον εθνικό δικαστικό τομέα και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος. Στο άρθρο 83 μιλάμε για διασυρωριακό έγκλημα. Благодаря, госпожо председател. Аз искам, може би, изненадващо за някои колеги да припомня какъв беше случая в навечер, с Албания в навечерието. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να θυμίσω την περίπτωση ε, της Αλβανίας, παραμονές άρσης θεώρηση των διαβα... διαβατηρίων. Και τι δεν ακούσαμε. Πανικός. Θα σηκωθούν όλοι οι Αλβανοί και θα έρθουν στην Ευρώπη. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα εσωτερικής πολιτικής στην Αλβανία. Δεν βλέπουμε κανένα τρομερό μεταναστευτικό κύμα. Δεν ήρθαν στην Ευρώπη όλοι οι Αλβανοί, απλούστατα, διότι υπάρχει οικονομική ανάπτυξη σχετικά ευσταθής σταθερή παρόλη την πολιτική κατάσταση. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι φόβοι, αγωνίες, ανησυχίες ότι θα μας κατακλείσουν οι Αλβανοί αποδείχθηκαν τελείως αβάσιμες. Είδαμε και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του Σέγγεν και θυμίζω ότι αυτός ο πανικός και αυτή η φόβη είναι κάτι που εμφανίζονται συχνά. Εντάξει, ενεχάρημε τον κύριο Κοέλιο για την ουσία της έκθεσής του, αλλά θα πρέπει να τον συγχαρούμε επίσης και μάλιστα να το βραβεύσουμε γιατί πραγματικά υπερασπίζεται την κοινή λογική και την ψυχραιμία. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε ε, καμία καταστροφή τώρα επειδή θα πει η Βουλγαρία και η Ρουμανία στο Σέγγεν. Πολύ δε περισσότερο που πρόσφατα τις τελευταίες μέρες προβλέψαμε μέτρα τα οποία θα αποδειχθούν οπωσδήποτε πολύ αποτελεσματικά και πολύ χρήσιμα. Συμφωνώ πολύ το στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους οργανισμούς αυτούς Eurojust, Europol κτλ. Με τρόπο όμως ε, σωστό, πλήρη, εμπεριστατωμένο, όχι αποσπασματικά αν θέλετε και 24 ώρες το 24ωρο. Διότι έτσι θα ε, διασκεδαστούν οι, ε, οι εικασίες. Θυμίζω ότι στην τελευταία έκθεση της Europol βλέπουμε περίεργες διαπιστώσεις για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που δεν βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά σοβαρές μελέτες ή αποδείξεις. Μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μελέτες, αλλά δεν βλέπουμε να αναφέρονται στην έκθεση αυτών των οργανισμών. Μια μεγάλη πόλη παραθαλάσσια στη βόρεια, στη Μαύρη Θάλασσα, συγγνώμη, χαρακτηρίζεται ως νέα πύλη εισόδου της αμερικανικής παρακαλώ κοκαίνης από την Ευρώπη. Αυτό πού το βρήκανε. Πώς το διαπιστώσαν. Είναι κανένα τρίγωνο, εκεί πρέπει να περάσει από τον εύξηνο πόντο. Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του εγκληματικού δικτύου. Όλα αυτά είναι εικασίες, ε, ανησυχούν τον κόσμο και είναι βάσιμα. Επίσης θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται λεπτομερέστατα και να ε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και να έχει και να ακούει και να πιάνει ό,τι συμβαίνει στο Σέγγεν. Πολύ συχνά εκθέσεις της Eurojust, της Europol και της Frontex είναι γραμμένες σε μια γλώσσα πάρα πολύ τεχνική, επαγγελματική και είναι πολύ δύσκολο ε, να ε, τις κατανοήσουμε, αλλά βλέπουμε ότι είναι συνταχνιακή η ψυχολογία που διέπει τους συντάκτες αυτών των εκθέσεων. Και θέλουν να επιδείξουν ε, είτε αλληλεγγύη με τους συναδέλφους τους των άλλων κρατών, είτε να τους στιγματίσουν ε, γιατί είναι απογοητευμένοι. Πώς να εξηγήσουμε, όταν έρχονται στη Βουλγαρία ε, οι υπάλληλοι της Frontex, της Europol, πάντα είναι πάρα πολύ ευγενείς, κάνουν δώρα, χαιρετούρες και μετά στο Συμβούλιο Υπουργών είναι οξύτατες οι κριτικές τους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να μην ε, ανεχόμαστε υποκειμενικές μελέτες γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Ευχαριστώ και ο, ο κύριος Μαρινέσκο θα είναι ο τελευταίος μας ομιλητής πριν ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας. Ο χώρος ε, Σέγγεν δεν προβλέπει μηχανισμούς επίγουσας ανάγκης για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ε, έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πλήττει την αξιοπιστία μας. Η εισαγωγή ελέγχων τώρα στα σύνορα είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεσπίσει ένα κράτος μέλος χωρίς να ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα μπορούσαμε να επανεισαγάγουμε ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα υπό έκτακτες συνθήκες και περιορισμένους στο χρόνο. Νομίζω ότι η επανεισαγωγή αυτών των μέτρων είναι ένα έκτακτο μέτρο και αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος μέλος δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις σε έξι μήνες. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο χώρος ε, Frontex και η ε, διαλειτουργικότητά του, όπως προβλέπετε. Η επανεισαγωγή ελέγχων είναι ένα μέτρο που τίθεται σε ισχύ αν το προτείνει η Κομισιόν, το Συμβούλιο ή πλειοψηφία κρατών μελών. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με εκπροσώπους των κρατών μελών και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζονται ε, χρηματοδοτικά μέτρα αντιστάθμισης εάν χρειαστεί να επανεισαχθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα και αυτό αφορά την όλη αξιολόγηση του χώρου Σέγγεν. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να εισαχθούν ήδη από τώρα στο κεκτημένο Σέγγεν. Τώρα δίνω το λόγο στον Κάρλος Κουέλιο για να, μας, για να συνοψίσει με βάση τα στοιχεία που άκουσε και να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι υπάρχουν κοινέ ανησυχίες, μιλάμε για διαφάνεια, για προστασία, μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι θέματα που μας βρίσκουν σύμφωνους. Δεύτερον, το ζήτημα είναι ότι όλοι έχουμε το ίδιο σημείο εκκίνησης. Το σημείο εκκίνησης ήταν να αναγνωρίσουμε ότι το παρόν σύστημα αξιολόγησης του κεκτημένου του Σέγγεν δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, διότι οι αναλύσεις μεταξύ ομοτήμων οδηγούν σε μία διαδικασία όπου το ένα κράτος μέλος δικαιολογεί το άλλο. Δηλαδή το ένα χέρι είναι βιτάλο. Μιλάμε για πιο λιγότερα επιβαρημένα μάλλον κριτήρια κατά τη στιγμή της ανάλυσης λιγότερες επιβαρύνσεις και δεν υπάρχουν επιτόπιες συνέπειες υπό το παρόν σύστημα αξιολόγησης του ΣΕΝΚΕ, με εξαίρεση τις υποψήφιες χώρες. Και στην Επίτροπη ΛΥΜΠΕ πολύ συχνά είπαμε ότι δεν δεχόμαστε δίπλα δύο μέτρα και σταθμά, δηλαδή άλλο σύστημα για τις χώρες που έχουν ενταχθεί και άλλο για τις υποψήφιες χώρες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα με επικεφαλή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα διαχειρίζεται το σύστημα. Ορισμένοι συνάδελφοι το προανέφεραν, γιατί μιλάμε για αμοιβαία εμπιστοσύνη Οι εμπειρογνώμονες, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες λοιπόν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες. Μας ενδιαφέρει μία ευρωπαϊκή προσέγγιση με τη συμμετοχή των κρατών μελών. Και αν διαμορφώσουμε το σύστημα κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα φτάσουμε σε έναν πολύ καλό μηχανισμό αξιολόγησης. Ορισμένοι συνάδελφοι μίλησαν για εισαγωγή νέων κριτηρίων. Σας είπα και προγενέστερα ότι μπορώ να δεχτώ τις ανησυχίες σε σχέση με τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Και θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Δηλαδή, σε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται μία στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα τη στιγμή που μπορούν να υποσκάψουν και να υποβαθμίσουν το παρόν σύστημα. Σε αυτό το κείμενο όμως νομικής εμβέλειας δεν μπορούμε να κινηθούμε πέραν αυτού διότι δεν διαθέτουμε νομική βάση. Ένα άλλο ζήτημα είναι να γνωρίσουμε και να αποφασίσουμε κατά πόσο στη νομική βάση του κεκτημένου του Σέγγεν θα πρέπει να γίνει μία διεύρυνση. Και μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε πρόταση των συναδέλφων για να διευρύνουμε τα κριτήρια αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το συγκεκριμένο μέσον. Δεν διαθέτουμε νομική βάση. Μπορούμε μόνο να αναφερθούμε στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, εάν μιλάμε για θέματα που υποβαθμίζουν το Σέγγεν. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τομείς όπως τα ναρκώτικα και την εγκληματικότητα όπου υπάρχει και διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτούς τους τομείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως προς τις τροπολογίες, δηλαδή Μακοβέη, Σάρα Λάντφορτ και Τίμωθη Κίρκοπ, γιατί πρέπει σε πρώτη φάση να εντάξουμε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα σε αυτό το νομικό κείμενο, έτσι ώστε να τα εντάξουμε στο προϋπάρχον και εκτιμένο και μετά να το διευρύνουμε σε ένα άλλο κείμενο με την εισαγωγή νέων κριτηρίων. Τέλος. Α, συγγνώμη, θα ήθελα να πω στη Μαρία το εξής. Όταν μιλάμε για μερικούς ελέγχους, τι εννοούμε. Ένας μηχανισμός αξιολόγησης σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε μία χώρα, όχι μόνο, όχι σε όλες. Και όταν μιλώ για συγκεκριμένα σύνορα, μιλώ για, ε, για τα σύνορα, για συγκεκριμένα σύνορα ή για μία χιλιομετρική απόσταση. Αυτό αφορά τα ε, σύνορα ε, από στερεάς, από θαλάσσης ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, εάν ότι πολλές φορές σε χώρες υπάρχει πολύ καλός έλεγχος και ασφάλεια στα, ως προς τα εναέρια σύνορα και τα ε, σύνορα από, από τη στεριά, αλλά όχι από τη θάλασσα. Γι' αυτό που, έχει, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πού έγκυται το πρόβλημα, εάν υπάρχει σε κάποια χώρα. ως προς την επανεισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε ένα πολύ καλό μηχανισμό αξιολόγησης με την ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με μεγάλη διαφάνεια σε επίπεδο κρατών μελών. Όταν αναγνωρίσουμε λοιπόν το πρόβλημα, τι πρέπει να γίνει. Και εδώ έχω υποβάλει μια τροπολογία. Εάν εντοπιστεί ένα πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και η πρώτη μας αντίδραση θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε το εν λόγω κράτος μέλος να επιλύσει το πρόβλημα με τη Frontex, με τα ευρωπαϊκά μέσα που διαθέτουμε. Τι θα κάνουμε όμως αν ε, εμένει το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε, θα ε, ε, εθελοτυφλούμε, θα λέμε ότι εντάξει καταβάλαμε προσπάθειες, δεν έγινε τίποτα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, ασφάλειας στα ενδοκινοτικά σύνορα και γι' αυτό θα πρέπει να προβληθούν κυρώσεις. Ας μην δραματοποιούμε. Αυτή τη στιγμή κάθε κράτος μέλος από μόνο του μπορεί να επανεισαγάγει ελέγχους στα σύνορά του. Εμείς ε, ζητούμε να υπάρχει μια συλλογική απόφαση. Εάν ένα κράτος μέλος επανεισαγάγει ελέγχου στα εσωτερικά του σύνορα, τότε γιατί να μιλάβουν την ίδια απόφαση τα άλλα κράτη-μέλη. Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα με συγκεκριμένα σύνορα και το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, η Frontex δεν αρκούσε. Τα ευρωπαϊκά μέσα δεν αρκούσαν για να βοηθήσουμε το κράτος μέλος τότε θα πρέπει να ληφθεί μια άλλη απόφαση. Να πούμε δηλαδή ότι θα επανεισαγάγουμε ελέγχου στα σύνορα, διότι όλα τα άλλα μέσα δεν ήταν αποδοτικά. ως προς την, ε, τους ελέγχους στα εξωτερικά δηλαδή σύνορα. Βεβαίως πρόκειται για ένα μέτρο που είναι το τελευταίο στην κλίμακα. Είναι ένας μηχανισμός αναχέτησης έτσι ώστε να αποφύγουμε μεγαλύτερα προβλήματα και θα πρέπει να είναι μία διαδικασία μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου. Απόφαση δηλαδή του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε όλα τα θεσμικά ε, όργανα να εμπλακούν. Κατά την άποψή μου, εάν δεν επιτύχουν έχουμε να συγκροτήσουμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης με ευρωπαϊκή προσέγγιση, συμμετοχή κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με αυτή τη συγκεκριμένη ιδέα, με αυτή τη συγκεκριμένη βάση θα, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχει κακή αξιολόγηση, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Διαφορετικά δεν θα βρούμε μία καλή λύση, δεν θα ανταποκριθούμε στην εντολή μας κύριε Πρόεδρε. Και κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γνωμοδότησή της. Συμμερίζομαι τα περισσότερα σχόλια που ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως μερικές τροπολογίες προχωρούν αρκετά μακριά, αλλά νομίζω ότι αποτελούν μια καλή βάση εργασίας και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβασμό μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Τώρα προς το Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι η Προεδρία πρέπει να μας αναφέρει την άποψη του Συμβουλίου. Είμαι αρκετά απογοητευμένος από το Συμβούλιο. Εάν κατάλαβα καλά, σταμάτησαν ε, ως προς τη νομική βάση και δεν θα συζητήσει τίποτα άλλο το Συμβούλιο μέχρι ότου ληφθεί μία απόφαση ως προς τη νομική βάση. Θα ήθελα να πω στο Συμβούλιο ότι αν αποζητούν να αλλάξουν τη νομική βάση, νομίζω ότι κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί οποιαδήποτε νέα νομική βάση για το μηχανισμό αξιολόγησης του κεκτημένου του Σέγγεν θα πρέπει να αποφασιστεί με τη συναπόφαση. Δεν υπάρχει άλλη νομική βάση. Θα πρέπει να είσαστε υπόλογοι στα κράτη-μέλη για τη νέα μορφή διακυβέρνησης και δεν δημιουργείται το καλύτερο δυνατό κλίμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία συναπόφασης με βάση την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν νομίζω ότι ε, είσαστε πιστοί όπως ορίζουν οι συνθήκες. Δηλαδή, αφού αρχίσει η νομοθετική διαδικασία, να αλλάξετε τη νομική βάση έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μην μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία συναπόφασης. Θα ήθελα να πω στο Συμβούλιο ότι ούτε σε νομικό ούτε σε πολιτικό επίπεδο θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα δοθεί απάντηση. Εάν το Συμβούλιο θέλει λοιπόν να ακολουθήσει αυτή την οδό, τότε θα λάβει μια στεναρή ανταπάντηση από εμάς. Αυτή είναι ε, μια πολύ άμεση απάντηση σε σχέση με τα αρνητικά αυτά βήματα που έλαβε το Συμβούλιο. Ε, ευχαριστούμε Κάρλο. Ήταν ε, σαφές. Σίγουρα θα ζητήσουμε μια παρουσίαση από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προβλέπετε να ακούσουμε τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας στην επόμενη μας συνεδρίαση που θα γίνει 12 και 13 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στη συζήτηση και περάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας που προβλέπει συζήτηση σχετικά με τη ΕΠΟΛ, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Η συζήτηση αυτή ε, λαμβάνει η χώρα μετά την άρνηση χορήγηση απαλλαγής της ΕΠΟΛ για τον προϋπολογισμό του 2009 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να, εξετάσουμε, να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Γι' αυτό και ε, προσκαλέσαμε τον Διευθυντή της ΕΠΟΛ, τον κύριο Μπάμφη, για να λάβει μέρος σε αυτήν την απογευματινή συζήτηση και πριν του δώσω το λόγο να σας υπενθυμίσω ότι είναι ο νέος διευθυντής της ΕΠΟΛ και από ό,τι φαίνεται έχουν λάβει χώρα ρηξικέλευτες αλλαγές ό,τι αφορά την ε, ηγεσία και τον τρόπο διοίκησης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Πριν ε, του δώσω το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, αν υπάρχουν τις απορίες τους, ώστε μετά να ακούσουμε τον κύριο Μπάμφη, τον διευθυντή της ΕΠΟΛ, που θα μας ενημερώσει για τις ε, δραστηριότητες και τις εξελίξεις στην, αστυνομία, στην Αστυνομική Ακαδημία. Η κυρία Ματιέ ζήτησε το λόγο. Ο άλλος συνάδελφος θέλει να θέσει ερωτήσει. Κύριε Ματιέ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας σήμερα μετά από την χορήγηση άρνησης απαλλαγής και συνεχίζοντας το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τη φορά την, τον έλεγχο του προπολογισμού. Έχουμε αρνηθεί την χορήγηση απαλλαγή στη ΕΠΟΛ για το 2008 και είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χορήγησε απαλλαγή σε έναν οργανισμό. Γι' αυτό και εξετάζουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας ε, με τα Διευθυντή και τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Θα ήθελα να σας επιθυμήσω ότι το μεταξύ ε, διορίστηκε νέος διευθυντής στις ΕΠΟΛ και δεν ευθύνεται ο κύριος Μπάμφη για την άρνηση χορήγησης της απαλλαγής γιατί αφορούσε το 2008 και, αυτός διορίστηκε, και εκείνος διορίστηκε αργότερα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας είναι να συμβάλλει στην επιμόρφωση των υψηλόβαθμων αξιωματικών της αστυνομία στην Ευρώπη και στον κόσμο και ταυτόχρονα η ενίσχυση του Σέγγεν ε, μας ε, οδηγεί στην ανάγκη πολύ πιο κατερτισμένου προσωπικού στην αστυνομία σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αν ε, η ΣΕΠΟΛ μπορεί να επιτελέσει το έργο της. Το 2010 είχε λιγότερο από 23 μέλη προσωπικό. Είναι ένας πολύ μικρός οργανισμός. Ουσιαστικά είναι σαν ε, μια γραμματεία ενός δικτύου υπαλλήλων που είναι ε, διασκορπισμένη σε διάφορα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γραμματεία βρίσκεται στο Μπράμψη, 70 χιλιόμετρα νοτίως του Λονδίνου, σε μια δυσπρόσιτη πόλη που δεν είναι καθόλου ελκυστική για να προσλάβει ε, ειδικευμένο προσωπικό. Και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, είχατε πέρυσι 45.000 ευρώ μόνο για ταξί. Θα μας ε, ενημερώσετε πιο διεξοδικά. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπερμεγέθεση σε σχέση με το μέγεθος της ΣΕΠΟΛ και αυτό αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο το, τον τρόπο λειτουργίας της. Και μάλιστα στο Διοικητικό Συμβουλίο τα κράτη-μέλη ε, εκπροσωπούνται από ένα ως τέσσερις εκπροσώπους, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομική Ακαδημίας. Προτείνεται τώρα να περιοριστεί σε ε, δύο μέλη κάθε εθνική αντιπροσωπεία, γιατί πιστεύουμε ότι αρκούν δύο εκπρόσωποι από κάθε κράτο, όπω και για άλλου οργανισμού. Έτσι θα μπορούσαμε να ελαφρύνουμε κάπως το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να μπορέσει η Ακαδημία αυτή να επικεντρωθεί στο βασικό της έργο. Σε ό,τι αφορά την έδρα της γραμματείας, τον ε, τόπο στον οποίο βρίσκεται. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί να μην μεταφερθεί η γραμματεία στις Βρυξέλλες, όπου δρεύει και ο Λάφη, στη Χάγη γιατί νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη στρατηγική, στρατηγικό συντονισμό και συνεργασία. Κύριε Διευθυντά, σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητώ το έργο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και την ανάγκη ύπαρξής της. Για μας είναι πολύ σημαντική. Ο οργανισμός σας είναι σημαντικός, ε, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη μορφή που έχει σήμερα. Βέβαια και εσείς καταθέσατε προτάσεις. Γνωρίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και άλλες προτάσεις. Πάντως, προσωπικά πιστεύω ότι η συγχώνευση της ΣΕΠΟΛ με την Ευρωπόλ δεν στέκει προτείνω να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, να μεταφερθεί η έδρα της. Γιατί στο Μπραμσίμ, εκεί 70 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, δεν είναι σωστή έδρα, ούτε λειτουργική για το έργο της ΕΠΟΛ. Ξέρω ότι καταβάλλατε τεράστιες προσπάθειες για να διαγράψετε κατά κάποιο τρόπο το παρελθόν, αλλά θεωρώ ότι για μας, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά και για την κατάρτιση των αστυνομικών, απαιτείται και ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και μετάθεση της έδρας της. Σας εύχομαι καλό κουράγιο και καλή τύχη στο έργο σας, κύριε Διευθυντά. Ε, Μόλις ε, βλέπω ότι ζήτησε το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρέμβει και μετά θα δώσω το λόγο στο Διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αν νόμιζα ότι δεν θα μιλούσα πρώτος εγώ, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα της αναθεώρησης της νομικής βάσης ε, και κατάστασης της Αστυνομικής Ακαδημίας προβλέπεται προς το παρόν για το 2013. Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή για την αναδιατύπωση, όπως είπαμε, της νομικής βάσης ε, της Αστυνομική Ακαδημία μέχρι τότε, το 2013. Δεν αποκλείεται να γίνει και νωρίτερα όμως. Και δεν σας κρύβω ότι μας απασχολεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γίνει νωρίτερα. Ζητήσαμε αξιολόγηση η οποία αναμένεται να κατατεθεί μέχρι ε, το καλοκαίρι του 2012 θα ερήνουν αυτά που λέγει η συγγήτρια ότι έχει και ρόλο ε, η ΣΕΠΟΛ και χρήσιμο δηλαδή και πάγιο και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μαθαίνω από τις υπηρεσίες επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως ανέφεραν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΠΟΛ, έχει αθωωθεί η αστυνομική ακαδημία ως προς κατηγορίες θεωρούν ότι είναι ένας οργανισμός ε, με υγιή πλέον οικονομική διαχείριση που είναι στο μέσο όρο των υπολείπων, να μην πω και άνω του μετρίου. θα ήθελα να ε, συγχαρώ και τον κύριο Δευθυντή για τα καθήκοντα που ασκεί από τότε που ανέλαβε. Η Σέπολη Αστυνομική Ακαδημία πρέπει να εκπαιδεύει μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ερχών Επιβολής της Τάξης. Αυτό το ζητάει άλλωστε το πρόγραμμα της Οκόλμης. Έχει ένα ρόλο πολύ ενδιαφέροντα, όσο και σημαντικό να διαδραματίσει το μέλλον και τώρα που έχει λύσει τα διοικητικά και τα οικονομικά της προβλήματα, είναι ακριβώς η στιγμή να αρχίσει να σκέφτεται τι πολιτικές χρειάζεται για ε, να εκπαιδεύει ε, στο μέλλον ε, στελέχη των αρχών επιβολής της τάξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλοί οργανισμοί και τα μέσα, αλλά είναι πολύ κρίσιμο να τα γνωρίζουν οι αποδέκτες αυτά τα όργανα για να τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Υπάρχει και πρόβλημα γνώσης και πρόβλημα ε, εμπιστοσύνης. Δεν είναι περιφερειακό το ζήτημα αυτό, είναι σημαντικό και στην καρδιά του προβλήματος ή των προβλημάτων που να αντιμετωπίζει ο χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης αυτό τον καιρό. So, bearing all this in mind, uh, Αυτά. Λοιπόν, πώς ε, έχουν τα πράγματα σήμερα, τώρα που έχει ε, σταθεί στα πόδια της η ε, ΣΥΠΟΛ, ο οργανισμός αυτός, που έχει επαρκή και χρηστή και ορθή διαχείριση. Ε, τώρα πρέπει να κάνουμε εικασίες για το αν θα μπορέσει να συγχωνευτεί με την Ευρωπόλ, με όλα τα συμπαραμαρτούντα και τις λειτουργίες και τα προβλήματα που θα ε, απορρεύσουν. Το ερωτώ αυτό προς όλους σας. Δεν θα ήταν περίεργο τώρα που μπορούμε να συγχαρούμε τον οργανισμό αυτό για όλη τη δουλειά που έκανε. Πρέπει να ανατρέψουμε ε, τη διοικητική μηχανή ολόκληρη και να συγχωνευτεί με την Europol. Αφήστε που και η Europol δεν το θέλει. Και ακόμα και αν ήταν καλή ιδέα αυτή που πολύ τολμώ να αμφισβητήσω, θα πρέπει να γνωρίζει και το Κοινοβούλιο ότι τι σημαίνει ε, διάλυση ενός οργανισμού, ε, κατάργησή του. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εάν πάρουμε αυτή την οδό, ε, θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Ακόμα και αν συμφωνήσουν τα 27 κράτη-μέλη, που δεν νομίζω ποτέ να συμφωνήσουν και τα 27, δεν είναι υπόθεση μηνών, μπορεί να είναι υπόθεση ετών αυτό. Και νομίζω ότι πιο χρήσιμο θα ήταν να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη, ε, στην υπεράσπιση και στην ενίσχυση της ΥΠΟΛ ε, για να μπορέσει στο μέλλον να κάνει σωστά τη δουλειά της και να εκπαιδεύει ε, τα στελέχη που χρειάζεται. Υπάρχει ένα σημείο που διαφωνώ με την συγγετρία, αν μου επιτρέπετε. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μου δίνει η γραμματεία της ΣΥΠΟΛ, δεν έχουν πρόβλημα προσλήψεων ε, προσωπικού ε, σήμερα στον οργανισμό. Τι σημαίνει αυτό. Καλά, το Μπράμσιν δεν είναι αγαπημένος προορισμός όλων ε, να ζήσουν. Μερικών τους αρέσει. Όχι όλων, αλλά δεν είναι πρόβλημα να βρουν ε, υπαλλήλου που θα πάνε να κατασταθούν εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι στις προσλήψει. Καλύπτουν όλες τις θέσεις τους ε, που ε, χειρεύουν και δεν νομίζω να είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν ξέρω, διαρωτώ. Αυτά για σήμερα και σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα συνάδελφο ζήτησε το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στο Διευθυντή, Μία συνάδελφος, μάλλον κυρία Μακοβέη. thank you very much. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα σε σχέση με την πρόταση συγχώνευσης της ΣΥΠΟΛ με τη Europol. Θα ήθελα να πω ότι η ετήσια έκθεση του 2009 σε εκείνη την έκθεση είχε προτείνει ή να αναλάβει αυτή τη διαδικασία εκπαίδευσης των υπαλλήλων. Άρα πρόκειται για μία θέση που προεπήρχε και θα ήθελα να πω ότι δεν θέλουμε να αποσταθεροποιήσουμε τον οργανισμό ή τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης. Θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματικότητα και ε, σωστή σχέση κόστους-οφελίας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πολιετές πλαίσιο 2011-2014 και θα ήθελα να επιμείνω και να πω ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στο πολιετές, κάτι το οποίο επικρίνεται από τον εσωτερικό έλεγχο ε, ορκωτών λογιστών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μιλάμε για αλλαγές στο διευθυντικό προσωπικό τώρα και δεν ξέρω κατά πόσο ε, μπορούμε να προσμένουμε μεγάλες αλλαγές. Θα ήθελα λοιπόν να μου μιλήσετε για την διαφάνεια στο ε, χρηματοδοτικό σχέδιο 2011-2014 και περιμένουμε και την έκθεση ετήσιας δραστηριότητας για το 2010 έτσι ώστε να δοθεί η απαλλαγή για το 2010. Τέλος, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και να λάβουμε υπόψη τη συγχώνευση, η οποία συζητιέται εδώ και μακρύ χρονικό διάστημα, γιατί να μην περιμένουμε πρώτα αποτελέσματα πριν προωθηθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα, όχι να έχουμε υψηλές δαπάνες και να δούμε τα διαρθρωτικά προβλήματα του, της Ακαδημίας. Δεν θα ήθελα να ε, ε, αναφερθώ στο γεωγραφικό χώρο. Είναι πολύ δύσκολο με βάση τα διοικητικά μέσα να αντιμετωπιστούν μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση. Αν δούμε την απαλλαγή για το 2009, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα λάθη ως προς τις διαδικασίες προμηθειών και σε ένα μικρό οργανισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι διορθώσεις. Νομίζω ότι η ΣΥΠΟΛ θα πρέπει να ενταχθεί στη Europol για να έχουμε εξοικονόμηση σε ευρεία κλίμακα. Να έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, καλύτερη συνεργασία, λιγότερες ε, δαπάνες και καλύτερο αντίκτυπο και συνεργασία με άλλους οργανισμούς όπως τη Eurojust που βρίσκεται που βρίσκεται στη Χάγη. Δεν μιλάμε για τους επόμενους μήνες, μιλάμε για την απαρχή μιας διαδικασίας. Και θα πρέπει να προβάλλουμε και τα σωστά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε Μόνικα. Τώρα αφού ακούσατε τις ε, διάφορες ε, ιδέες και επιχειρήματα, δίνω το λόγο στο Διευθυντή της ΣΥΠΟΛ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εργασία σας ε, σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ που προσήλθατε για απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Είναι η πρώτη φορά που έχω ε, λάβει μία πρόσκληση από την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι πέρσι το Φεβρουάριο όταν ανέλαβα τις εργασίες μου στο Bramshill, βρήκα ε, μία, ε, έλαβα μάλλον μία, αντιμετώπισα μία πολύ βαριά κληρονομιά. Είχα να ε, διαχειριστώ μία μεγάλη κρίση έτσι ώστε να τηρηθεί το γράμμα του νόμου και για να αναλάβω με επαγγελματισμό αυτό μου το έργο. Οι, δυσκολίες της Ακαδημίας δεν σχετίζονται με το μέγεθός της, αλλά επειδή δεν υπήρχε σωστή ε, ηγεσία. Και αυτό φαίνεται από τις επιτυχίες μέχρι τώρα. Πέρσι έπρεπε να αντιμετωπίσω και να διαχειριστώ ε, μία κατάσταση κρίσης και φέτος φαίνεται ότι ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Δυστυχώς χάσαμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρώ προσωπικά ότι αυτό αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες, τις υψηλότερες προτεραιότητες, δηλαδή να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη σας. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο εξής. Όλα τα πρόσωπα τα οποία δημιούργησαν δυσκολίες δεν είναι πλέον ενεργά μέλη. Έχω 37 συναδέλφους έχουμε 26 προσωρινούς συμβασιούχους δηλαδή και 10 και επιπροσθέτως 45 ε, μισθωτοί εργάζονται με βάση το δίκτυο της ΣΥΠΟΛ σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ακαδημία ε, είναι, ε, έχει μία ε, νόμιμη δραστηριότητα και διαφανή δραστηριότητα. Άρχισαν οι ελέγχοι από πέρσι από, τον, από το ελεγκτικό συνέδριο τον Οκτώβριο του 2010. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν βρήκε καμία παρατυπία και παράλληλα ο εσωτερικός έλεγχος με βάση το πολιετές ε, ε, πρόγραμμα, δημοσιονομικό πρόγραμμα, ε, προέβησε ελέγχους μέσα στα πλαίσια του δεκαετού σχεδίου. Ήθελα λοιπόν να υπάρχει πλήρης διαφάνεια όλων, ολόκληρης της λειτουργίας τη ΣΥΠΟΛ, γι' αυτό και σας υπέβαλα αυτή την έκθεση αργότερα. Φέτος, με βάση το δικό σας ε, αίτημα, το ελεγκτικό συνέδριο διενέργησε ε, δύο ελέγχους μέσα στα πλαίσια του δεκαετούς δημοσιονομικού προγράμματος και φτάσανε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν παρατυπίες στο δεκαετές σχέδιο. Το Μάιο, επιπροσθέτως, το ελεγκτικό συνέδριο διενέργησε έναν νέο έλεγχο για τους λογαριασμούς μας από το 2010, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και προμήθειες. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ακαδημία έλαβε άριστα σε όλους τους τομείς δεν υπήρξαν σχόλια, αρνητικά σχόλια ή επικρίσεις σε σχέση με τα αποτελέσματά μας. Ε, δηλαδή, πληρούμε όλες τις νομικές προϋποθέσεις. Επίσης, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αναθεώρησε την ιστοσελίδα της Ακαδημίας και εκτίμησε, αξιολόγησε τη διαφάνειά μας και έφτασε στο συμπέρασμα ότι στο σελίδα της Ακαδημίας είναι διαφανής, φιλική προς το χρήστη και δίνει όλες τις πληροφορίες. Υπάρχουν βεβαίως οι υψηλές προσδοκίες να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, γι' αυτό ακριβώς δημοσιεύσαμε και τον προϋπολογισμό μας και ως προς τις τρέχουσες προμήθειες αλλά και ως προς τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλες μας τις δραστηριότητες από την ιστοσελίδα. Με βάση το δεκαετές σχέδιο και την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ακαδημίας η αξιολόγηση για την πενταετία έληξε και υποβλήθηκε στις ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια υπήρξαν επτά συστέσεις και μπορώ να σας πω ότι όλες οι ομάδες εργασίας για την εφαρμογή του νόμου έλαβαν υπόψη τα, όλα τα δεδομένα με βάση και το άρθρο 36 του κανονισμού. Ε, άρα γνωστοποιήθηκε η αξιολόγηση του πενταετού σχεδίου και οι επτά συστάσεις. Με λύπη μου θα πρέπει να αναφέρω ότι οι διοικητικές ε, δυσκολίες δυστυχώς επισκίασαν τις, ε, την καλή αποτελεσματικότητα και την απόδοση του δικτύου μας. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το πραγματικό μας, το ουσιαστικό έργο. Σε σχέση με τη νέα εγκατάσταση, βεβαίως το θέμα αυτό είναι καθαρά πολιτικό, δηλαδή η έδρα της ΣΥΠΟΛ βρίσκεται σε μία απόφαση του Συμβουλίου. Γι' αυτό οι υπουργοί θα αποφασίσουν για ενδεχομένη αλλαγή. Θα πρέπει όμως να υποθεί το εξής. Δεν ισχύει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών θέσεων εξαιτία της τοποθεσίας. Από πέρσι το Φεβρουάριο λάβαμε 600 αιτήσει. Υπάρχουν δηλαδή 20 υποψήφοι αναθέσει και πρόσφατα για μία θέση λάβαμε 90 αιτήσει. Μπορέσαμε να διορίσουμε τους υποψήφιους και υπάρχει και κατάλογος επιλαχόντων για να έχουμε και τους καταλληλότερους για τις σωστές ε, θέσεις. Ως προς το Συμβούλιο και τις Επιτροπές έχουμε αλλάξει τα σχέδιά μας και μπορώ να σας πω ότι η συμβουλευτική φύση και η διαβούλευση με το ελεγκτικό συνέδριο ή ο εσωτερικός λογιστικός έλεγχος υπάρχει. Καταλαβαίνω τις επικρίσεις σας, κατανοώ την απογοήτευση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί κάθε χρόνο ακούγατε ότι κάτι θα κάναμε, ε, και δεν κάναμε τίποτα. Αυτή τη φορά όμως τα καταφέραμε. Νομίζω ότι επεκτάθηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε και μπορώ να σας δώσω απαντήσεις αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάνφη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ε, λεπτομερείς πληροφορίες αυτές. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Εάν όχι, να σας συγχαρούμε για την εργασία που επιτελέσατε σε μία τόσο σύντομη χρονικό, χρονική περίοδο και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ συνάδελφε, ήταν το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, άρα τελειώνουμε στην ώρα μας. Λύεται η συνεδρίαση, η προσεχή συνεδρίαση της ΛΥΠΕ θα γίνει στις 12 και Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.